Κύριε Präsident. και κύριοι, καλημέρα σας. Έρχεται συνέδρια. Θα ήθελα να σα ενημερώσω ότι δεν έχει κατατεθεί κανένα αίτημα για ψηφοφορία για, το, για την πρόταση αυτή τη στιγμή και έτσι θα εγκριθεί όπως έχει. Προχωρούμε στη συζήτηση. Προετοιμασία για τι συνεδρίε του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και να το λόγο στον κύριο Λετσκεβίτσιου. Uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αξιότιμοι Ευρωβουλευτές, Πρόεδρε Τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Πολύ χαίρομαι που σήμερα το πρωί συμμετέχω στη συζήτηση αυτή σε σχέση με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τη επόμενη εβδομάδα. Υπάρχουν πολλά πράγματα στην ημερήσια διάταξη, μεγάλο εύρο θεμάτων που έχουν να κάνουν με την άμυνα, την Οικονομική και Νομισματική Ένωση, την Οικονομική και